So, welcome. Καλώς ορίσατε, συνάδελφοι από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Κυρίσω την έναρξη της κοινή συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΟΝ και της Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό. Ζίγκφριντ, έχετε το λόγο ως πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα και από εμά τους συναδέλφους της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Έχουμε κοινή συνεδρίαση των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μπράιαν Χαΐς για τα θερμά του λόγια. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της κοινή επιτροπής μας. Εάν όχι, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Δεύτερον, μπορούμε να εγκρίνουμε, εγκρίνουμε τα πρακτικά της 22ης Δευτέρας Οκτωβρίου του 18, της 25, της 5ης Οκτωβρίου, της 26ης και 27ης Νοεμβρίου του 2018 και της 3ης Δεκεμβρίου του 2018 επίσης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτά τα πρακτικά, θεωρείται ότι εγκρίνονται. Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις από πλευράς ε, Προεδρίας. Και γι' αυτό προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η ψηφοφορία για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Έχουμε δύο συναδέλφους ε, που έχουν ε, ε, δουλέψει ως εισηγητές, ε, κυρίως ο Μάνκα και Σίλβα Περέιρα, πάνω από 200 τροπολογίες και οι δύο εισηγητές έκαναν μια πολύ καλή συντονισμένη δουλειά και έχουν καταλήξει σε συμβιβαστικές τροπολογίες, οι οποίες έγιναν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους τρεις σκιώδες εισηγητές σε τρεις, με τους σκιώδες εισηγητές σε τρεις συνεδριάσεις που ήταν αρκετά μακροχρόνιες. Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία να δούμε αν λειτουργεί σωστά το σύστημα, παρακαλώ. Πέρας της ε, δοκιμαστικής ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε λοιπόν τώρα την ε, κανονική ψηφοφορία. Τροπολογία 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 1, 2, 3 και 4 ταυτόσημες ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική Γ. Σ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ. Κατά. Αποχές Ας το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 102 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική δέλτα. Με προφορική τροπολογία από την ΚΟΕ που προσθέτει το εξής κείμενο στο τέλος της συμβαστικής δέλτα ως μέρος μίας νέας πιο αηφόρου συμπεριληπτικής και δημοκρατικής οικονομικής διακυβέρνησης. Ως μέρος ενός τέτοιου νέου πλαισίου δηλαδή. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία, κύριε Γκλίντς. Εφτά μέλη πρέπει να έχουν αντιρρήσεις για να μην τη θέσουμε σε ψηφοφορία. Ποιος έχει αντιρρήσει. Ένας, δύο, τρεις. Σηκωθείτε παρακαλώ εσείς που είστε κατά. Ναι, είναι πάνω από 7. Άρα η προφορική τροπολογία δεν τίθεται προς ψήφιση. Άρα δεν την ψηφίζουμε και ψηφίζουμε τη συμβαστική δέλτα ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη τροπολογία 132 από τον κύριο Σβέν Κίγκολτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 134. Επίσης με προφορική τροπολογία από τους συναδέλφους των Πρασίνων και διαβάζω την προφορική τροπολογία. Υπογραμμίζει ότι σε μακροχρόνια βάση ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμβάλλει ε, κατά ένα μερίδιο στους πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για να δώσει στο Κοινοβούλιο την πολιτική ισχύ να ασκούν τα δικαιώματα ελέγχου του προπολογισμού ε, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής. είναι κατά να σταθεί όρθιος παρακαλώ. Ο οποίος δεν θέλει προφορική αυτή η τροπολογία να τεθεί προς ψήφιση. Βλέπω ότι είστε πάνω από 7, άρα δεν ε, τίθεται προς ψήφιση η προφορική τροπολογία. Αυτό σημαίνει ότι ψηφίζουμε την τροπολογία 134 όσα έχει χωρίς την προφορική της τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 158 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά Πρέπει να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε δια της ηλεκτρονικής οδού την τροπολογία 162. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Εγώ ψήφισα λάθος, γι' αυτό είπα, έβγαλα αυτό το επιφώνημα λάθος. Κοίταζα τον κατάλογο ψηφοφορίας της Προεδρίας και όχι τον κατάλογο ψηφοφορία τη πολιτική μου ομάδα. Δεν είχε αυτό τελικά σημασία, κάτι το οποίο δείχνει πόσο μικρή σημασία έχει ο πρόεδρο. Τέλο πάντων, πάμε στην 182 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 182 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Σαφέστατα απορρίπτεται. Συμβιβαστική H. Ήτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά πρέπει να επαληθεύσουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 211 πέρας Απορρίφθηκε. 223 υπέρ. Υπέρ 223 κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 237 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Ε, η 5 υπέρ κατά. Αποχές Νομίζω ότι εκρίνεται η αιτιολογική αναφορά υπαριθμών 5, το citation 5. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 6. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι το ίδιο. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 6 για της ηλεκτρονικής οδού. Πέρασα. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Δύο ψήφοι διαφορά ήταν πριν. Η 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Η και 13 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμε. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ψηφίζουμε λοιπόν το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το αρχικό κείμενο 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άρα ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο για την 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά Πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 20 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 31. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική Β με προφορική τροπολογία από την ΚΟΕ, την οποία διαβάζω εκεί όπου ο συμπεριληπτικός διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με σεβασμό στις εθνικές ιδιαιτερότητες, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την απλούστευση θα διασφαλιστεί. Θα διασφαλιστούν όλα αυτά. Υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτή την προφορική τροπολογία. Βλέπω πως όχι, άρα τη θέτω πως προς ψήφιση. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβαστική Β χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική Β λοιπόν εγκρίθηκε ως έχει χωρίς την προφορική τροπολογία και επειδή εγκρίθηκε αυτή πάμε κατευθείαν στην τροπολογία 226 η οποία συμπεριλαμβάνει προφορική τροπολογία από τους συναδέλφους από τους σοσιαλιστές και δημοκρατικές και το διαβάζω. Πιστεύει ότι οποιαδήποτε προσωρινή ρύθμιση που έχει ε, συναυθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του νέου ESF δεν θα πρέπει να γίνεται κατανοητή ω σημάδι που αυξάνει την αυτονομία του Δευτέρου, όταν η ισχυρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι θα έπρεπε, καθώς προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχει ε, συμπεριληφθεί στη συνθήκη και ε, στην ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αυτή η προφορική τροπολογία, γι' αυτό και πρέπει να μην ψηφίσουμε ξεχωριστά την τροπολογία 2.26 γιατί εγκρίθηκε η συμβαστική Β και δεν εγκρίθηκε η προφορική τροπολογία. Γι' αυτό πάμε κατευθύνς αμέσως στην τροπολογία 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 41. Πέρασα. Απορρίπτεται όντως. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57. Τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 ψηφίστηκε ως μέρος του συμβιβασμού και γι' αυτό πάμε στο αρχικό κείμενο. Για αυτή την αιτιολογική σκέψη Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 116 Sven Giggold. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 117. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο για την παράγραφο 7, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 56 από την κυρία Τομά αποσύρεται. Γι' αυτό και προχωρούμε στη συμβιβαστική F. Την ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 133. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην 92. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πρέπει να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 92. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 92. Τώρα αναφορικά με τις γνωμοδοτήσεις και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων πρέπει να ψηφίσουμε την αιτιολογική σκέψη Δέλτα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται συνάδελφοι. Για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, εξωτερικών Συνταγματικών Θεμάτων έχουν όλα καλυφθεί και γι' αυτό ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 59 ψήφους υπέρ, 25 ψήφους κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια στους δύο εισηγητές, τους συναδέλφους Σίλβα Περέιρα και Μάνκα. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά την οποία ολοκλήρωσαν οι δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.